Η συμφωνία που ετοιμάζουν κυβέρνηση και δανειστές μπροστά στη Σύνοδο Κορφής οδηγεί στην Καρμανιόλα την εργατική λαϊκή οικογένεια στην Ελλάδα. Προβλέπει νέα αντιλαϊκά μέτρα, διατηρώντας τα σκληρά μέτρα των προηγούμενων κυβερνήσεων από το λεγόμενο σκίσιμο των μνημονίων που υποσχόταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ εισηγείται τώρα στους δανειστές νέο μνημόνιο για να εξυπηρετείτε στο ακέραιο το αβάσταχτο χρέος της πλουτοκρατίας που δεν οφείλει ο λαός. Με αυξήσεις στους έμεσους φόρους, ιδιωτικοποιήσεις, κατάργηση ασφαλιστικών δικαιωμάτων, αύξηση ασφαλιστικών εισφορών φαίνουν νέες αβάσταχτες απώλειες στο ήδη πετσοκομμένο λαϊκό εισόδημα το κομμουνιστικό κόμμα της ελλάδας καλεί το λαό χωρίς αναμονή να απορρίψει τους εκβιασμούς να απορρίψει τα κυβερνητικά καλέσματα για υποταγή στο ρεαλισμό του ευρωμονόδρομου και του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης που φέρνει την εξαθλίωση και τη φτώχεια να εναντιωθεί στη νέα αντιλαϊκή συμφωνία και να μπλοκάρει τα αντιλαϊκά μέτρα αρνούμενος το χρέος να απαιτήσει την κατάργηση των μνημονίων και την ανάκτηση όλων των απολειών στον δρόμο της πραγματικής ρήξης με την ευρωπαϊκή ένωση το κεφάλαιο και την εξουσία τους. Πριν να δώσω το λόγο στον πρώτο αντιπρόεδρο της Επιτροπής, την κύριο Τίμερμανς και την κυρία Καλίνγκα Λουκασέβικα. Έχω την χαρά να σας πω ότι μια αντιπροσωπεία του Ινδικού Κοινοβουλίου έχει πάρει θέση στου ε, στους Νεξώστη. Καλωσορίσατε λοιπόν ε, θερμά, σας καλωσορίζω. Guidata dall'onorevole Presidente eh, Sabah, η ηγέτη της αντιπροσωπής, ο, κύριο ο κύριος Δελότης, ο Μάτης Σμήτρα Μπάγιαν. Και στόχος είναι να ενισχυθούν οι δεσμοί ανάμεσα στα δυο μας κοινοβούλια. Οι επαφές ανάμεσα στα δύο κοινοβούλια γίνονται από το 1981 και η σημασία της Ινδίας για να αυξάνεται όλο ένα, όπως αποδεικνύεται και από τη στρατηγική Συμφωνία που ε, θεσπίστηκε το 2004 και η συνεργασία μας με την Ινδία έχει οδηγήσει σε μια σειρά επισκέψεων στη χώρα. Τα πιο τελευταία ήταν τον Μάρτιο